Καλημέρα σας όλοι. Ελπίζω να έχετε μαζί σας τις κάρτες ε, ψηφοφορίας. Θα ξεκινήσουμε με τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Παρακαλώ, βάλτε στα μηχανήματα. Η πρώτη ψηφοφορία σήμερα είναι μια ένσταση όσον αφορά το λασάρισμα στην αγορά ε, προϊόντων ε, τα οποία περιέχουν γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι. Ε, και μια άλλη για το γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο. ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, άρχεται ψηφοφορία and it's closed. Στις ψηφοφορίες εγκρίνεται. Η δεύτερη ψηφοφορία είναι και πάλι μια ένσταση όσον αφορά την έγκριση της εισαγωγής στην αγορά προϊόντων από αραβάστο GA21. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Now we move to a report by Madame Gardini on the... Μια έκθεση της κυρίας Γκαρντίνη, πρόταση, απόφαση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου τροποποίηση απόφασης του 2013 όσον αφορά το μηχανισμό προστασίας των πολιτών. Ε, τροπολογία υπαριθμών 32 επέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, Προπολογισμό 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, Προπολογισμό 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 14 υπέρ κατά γίνει ευαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. 15, Ρέτζι, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 100, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 103 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 109 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 101 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 102 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 18 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 20 υπέρ, κατά, δεν ξέρω τι κάνουν εδώ πράσινοι. Πάμε που το λέω, αλλά απορρίπτεται. Υπέρ παρόλα αυτά. Κατά. Κατά απορρίπτεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 112 Όχι, λέει πρόεδρος, 114 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται, Ρέτζι. Μα έχει εγκριθεί το 113, λέει πρόεδρος. Want Επαλήθευση για την 21. 113. Είχε εγκριθεί 113. Ωραία, ας γίνει επαλήθευση. 113. 113. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ, κατά, αποχές, ελκ, 116 είστε υπέρ, ωραία και πάλι υπέρ, 116, κατά, αποχές, επαλήθευση για την 116, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 114 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 119 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 120 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 121 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 133 υπέρ, κατά ε, λυπάμαι, επανάληψη, 133, υπέρ. Κατά, αποχές, επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 134 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ρέτζι 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ρέτζι 24 υπέρ, κατά αποχές επαλήθευση Ρέτζ 24 άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ρέτζ 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ρέτζ 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 137 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για την 137 άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 139 και 140 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 142 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ρέτζι 27 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πολλές σελίδες. Μετά. 219, 219 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Προπολογισμό 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, Προπολογισμό 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 221 μέχρι 227 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 224 υπέρ υπέρ για την 224 ψηφίζουμε κατά αποχές, επαλήθευση για τη 224 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 225 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύε 8 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 98 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 226 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ντεβε 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 228 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 229 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προπολογισμό 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 230 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 231 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 232 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 233 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ρέτζι 37 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 234 ΕΠΕΡ κατά. Επαλήθευση για τη 234, άρχεται η ψηφοφορία. Όχι, έχει απορριφθεί. Ε, απορρίφτεται μάλλον, συγγνώμη. 235 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 248 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 247 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 236 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 239 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 240 υπέρ, κατά, Κατά. Επαλήθευση για τη 240. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 241 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 242 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 243 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 245 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία από τον εισηγητή τη μου για το άρθρο 1, παράγραφος 1, ε, άρθρο 15. Υπέρ της προφορικής τροπολογίας. Κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 11. Υπέρ κατά. Όχι, καταπίπτει, έχει καταπέσει. 248 και 249 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 250 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 251 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για τη 251 άρχεται η ψηφοφορία Πέραση της ψηφοφορίας απορρίπτεται η 38 υπέρ, ε, της Ρέτζη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 252 επερ κατά αποχές απορρίπτεται. 253 επερ κατά αποχές εγκρίνεται. Προπολογισμός 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ κατά αποχές, επαλήθευση για την 1, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27. Καταπίπτει. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ρέτζι 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29. Υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Άρχεται. Αν σας είχα πει ότι δεν είχατε τους πράσινους, θα γελούσατε. Πέρας, εγκρίνεται. 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται.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 Ρέτζι 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 8 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Budget 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. απόχέ απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά. απόχέ απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε την 74. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 76. Α, θα σε ελέγξουμε, εντάξει. Την 75. Πέρας, απορρίπτεται. 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μπάτζετ 4. Α, όχι. 79 και μπάτζετ 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε την 80. Άρχεται. And Πέρας, απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 81 και ρέντζε 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 83. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 84. Υπέρ. Κατά αποχές, ας ελέγξουμε την 84. Άρχεται. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Εγκρίνεται. Δεύε 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 12 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε την 85. Άρχεται. Πέρας απορρίπτεται. 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε τον 89. Πέρας. Εγκρίνεται. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 91 έως 93 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 94 έως 96 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. And it's closed. Πέρας. Εγκρίνεται σε χαρητήρια. Τώρα θα περάσουμε σε μία γνωμοδότηση ιδία πρωτοβουλία η Ευρώπη σε κίνηση, θεματολόγια για το μέλλον της κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 περ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε την 56. Πέρασε. Απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 66 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 68 πάλι σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 72 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 73 υπέρ, κατά άποχες έγκρινεται. 74 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται. And it's closed. Πέρας. Έγκρινεται. Συγχαρητήρια. Αυτό ήταν υποδειγματική, ε, ε, υποδειγματικός κατάλογος ψηφοφορίας με πολλές συμβιβαστικές. Τώρα θα ψηφίσουμε για το σημείο 19 τη διαφανή και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων σε αναπτυσσόμενες χώρες ή περίπτωση των δασών. Έκθεση Κονέτσνα. Συμβιβαστική 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά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 Τέλος. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές <clears throat> έλεγχος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 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 49 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 53 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε. And it is Πέρας απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, συγγνώμη, 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 72 υπέρ κατά αποχές Ας ελέγξουμε την 72. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 7 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 75 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές. Το ECR τι κάνει. Είστε υπέρ. Εγκρίνεται τότε. 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Α, ας ελέξουμε την 80. Ήταν αυτή η 80, ωραία, η 81 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα, έκθεση Δαντά, πρόταση για κοινού κανόνε για ορισμένε συνδυασμένε εμπορευματικέ μεταφορέ ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ε, τροπολογία 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83, 84, 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, υπέρ, 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται κατά αποχές απορρίπτεται 93 ε, υπέρ κατά αποχές 24 ε, απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά ας ελέγξουμε Δεν ψηφίζετε όλοι. Κάποιος ξέχασε την κάρτα του. Εγκρίνεται πάντως. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 105 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές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 εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τον, το, έτσι νόμιζα, αλλά δεν είχα δει κανένα χέρι. 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ υπέρ κατά έλκα πέρ κατά τότε απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 63 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 6 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά. Αποχές όχι κατά. Στο κατά είμαστε. Ποιοι είναι κατά της 16 ε, 14, συγγνώμη, 14 εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι, απορρίπτεται, απορρίπτεται, συγγνώμη. 17 ε, υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, σε 77 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές ποιος είναι κατά Ας ελέγξουμε τη 19. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Εγκρίνατε. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε τις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η κοινή ε, δημόσια κρόαση με την Επιτροπή Γεωργίας για τις νέες τεχνικές αναπαραγωγής και είναι στην αίθουσα της Επιτροπής Γεωργίας πιο πέρα, εδώ στον ίδιο διάδρομο. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ. Καλά